Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Σα καλωσορίζω στην Συνέδριση τη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ε, προτείνω να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 1, έγκριση τη ημερησία διάταξη. Ε, μία διευκρίνηση σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση αύξησης του αριθμού των δικαστών στο ε, τροτοδικείο. Ο εισηγητής ε, αντικαθίσταται για λόγους εσωτερικής πολιτικής της Πορτογαλικής Αντιπροσωπείας. Ε, ο, το όνομα του αντικαταστάτη δεν μας έχει κοινοποιηθεί. Ελπίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο τις επόμενες μέρες. Εν πάση περιπτώσει το σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση ήταν ήδη διαθέσιμο. Αυτό είναι κάτι θετικό. Δυστυχώ δυστυχώς όμως μόνο στα πορτογαλικά. Η αγγλική μετάφραση θα είναι έτοιμη αύριο το πρωί. Οι άλλες γλωσσικές εκδοχές θα ακολουθήσουν. Ε, δεν πρέπει να κατηγορήσουμε την υπηρεσία μετάφρασης. Ε, το κείμενο ήταν στα πορτογαλικά, χειρόγραφο και μακροσκελές. Γι' αυτό το λόγο καθυστέρησαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μέση αδιάταξη υπάρχουν αντιρρήσεις, προτάσεις. Κανείς δεν ζητάει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Θα ήθελα να σα συζητήσω να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη συνεδρία τη 13η και 14η Ιουλίου, τα τελευταία πρακτικά που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρία μα, θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται. Επόμενο σημείο. Το θέμα της κυρίας Ντελβό. Παρακαλώ, κυρία Ντελβό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για το θέμα της ε, αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, απλοποίηση της διαδικασίας, κάτι που θα βοηθούσε πολύ τους πολίτες που μετακινούνται για να εργαστούν ή για να διαμείνουν σε άλλο κράτος μέλος. Δεν θα σας συνοψίσω όλο το ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σε πρώτη ανάγνωση την γνωμοδότηση, την ε, γνωμοδότηση του. Μετά το Συμβούλιο καθυστέρησε, αλλά υιοθέτησε κοινή θέση και τώρα βρισκόμαστε στον τριμερή διάλογο. Μία συνάντηση έλαβε χώρα τον Ιούλιο, πρώτη συνάντηση επαφής και η δεύτερη συναδρίαση θα λάβει χώρα την πέμπτη αυτή τη βδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε μια κοινή θέση με το Συμβούλιο. Να πούμε ότι τα προσκόμματα είναι καταρχήν το πεδίο εφαρμογή, γιατί το Κοινοβούλιο είχε διευρύνει το πεδίο εφαρμογή, το Συμβούλιο ε, το συρρήκνωσε, περιορίζοντάς το σε ε, έγγραφα που έχουν σχέση με την οικογενική κατάσταση, γέννηση, θάνατος, ε, ε γάμος, σχέση πατρότητας κλπ. Το Κοινοβούλιο ήθελε να συμπεριλάβει και έγγραφα που άπτονται στην πρώτη ανάγνωση ενώ είχε προτείνει το Κοινοβούλιο να περιλάβουμε και έγγραφα για την κοινωνική ασφάλιση, τα διπλώματα και η Κομισιόν στην δική της αρχική πρόταση είχε επίσης προβλέψει να περιληφθούν και έγγραφα που αφορούν τις επιχειρήσεις ε, και τον, το είδος της επιχείρησης. Ε, το Συμβούλιο συρρήκνουσε λοιπόν το πεδίο εφαρμογής και βρισκόμαστε σε συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεύτερον, συζητούμε τα επικυρωμένα αντίγραφα το Κοινοβούλιο είχε προτείνει αν ένας ε, πολίτης υποβάλει μία δική του μετάφραση σε ένα δημοσιογράφο αυτή η μετάφραση να γίνεται δεκτή από το κράτος μέλος και αν υπάρχει κάποια αμφιβολία για την ακρίβεια της μετάφρασης τότε το, το κράτος μέλος να μπορεί να ζητά ε, ένα επικυρωμένο ε, αντίγραφο ε, ή ε, να προσφύγει στο IMI, το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών, που είναι η πλατφόρμα που ενώνει τις εθνικές διοικήσεις. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί με αυτό. Ορισμένες αντιπροσωπείες ε, αμφιβάλλουν για τη σκοπιμότητα της συμπερίληψης αυτής της διευκόλυνσης για τους πολίτες. Τρίτο σημείο, πρόσκομα, εμείς επιμένουμε ότι επιθυμούμε στην οδηγία να καταστεί σαφές πως τα κράτη-μέλη, οι υπηρεσίες των κρατών μελών έχουν την υποχρέωση να ε, ενημερώνουν τους ε, πολίτες ότι δεν έχουν πλέον ανάγκη επισημείωσης από στυλ. Στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται. Ε, αυτή τη στιγμή αυτή η υποχρέωση υπάρχει μόνο στην αιτιολική έκθεση αλλά όχι στο κείμενο. Επίσης θέλουμε ε, το κόστος ε, ενός πολύγλωσσου εγγράφου να μην το εντύπου, συγγνώμη, ε, να μην μπορεί να ξεπερνάει για το κόστος του πρωτότυπου εντύπου. Ε, αν δηλαδή ο πολίτης ζητήσει ένα πολύγλωσσο έντυπο, το κράτος μέρος μπορεί να ε, εισπράξει ένα ποσό για αυτό, αλλά αυτό το ποσό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ποσό το οποίο θα ε, εισέπρατε το κράτος για την πώληση ενός μονόγλωσσου εντύπου. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητούμε ε, είναι το θέμα των συμβολογραφικών πράξεων. Εδώ έχουμε ένα θέμα ορολογίας, ε, αφενός και αφετέρου, όπως γνωρίζετε. Όπως γνωρίζετε υπάρχει και η Σύμβαση της Χάγης που ε, ρυθμίζει τα, της, τα θέματα της επισημειώσεως. Το Συμβούλιο υιοθέτησε ε, την ορολογία της Σύμβασης της Χάγης ε, που όμως δεν συμπίπτει με την ορολογία που χρησιμοποιείται στα ευρωπαϊκά κείμενα και αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Αυτά είναι τα θέματα που συζητούμε στο τριμερή διάλογο. Ελπίζω να τελειώσουμε γρήγορα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο δυνατό περισσότερα. Απ' την άλλη μεριά όμως θα έλεγα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία μεταξύ των υπηρεσιών των κρατών μελών. Κανένα κράτος μέλος δεν εμπιστεύεται ε, έγγραφα, εύκολα έγγραφα ενός άλλου κράτους μέλους. Οπότε, αν τα καταφέρουμε να δημιουργηθεί ένα σύστημα ε, με βάση το οποίο τα κράτη-μέλη θα επικοινωνούν μεταξύ τους και θα δέχονται έστω και ένα μικρό αριθμό εγγράφων άλλου κράτους μέλους, θα είναι ένα πρώτο βήμα. Γιατί έτσι θα εδρεωθεί και μια σχετική εμπιστοσύνη, μια σχετική συνήθεια ε, ανταλλαγή πληροφοριών και διαβούλευσης Οπότε είμαι πρόθυμη να δείξω συμβιβαστικό πνεύμα αν συμφωνήσετε μαζί μου βέβαια. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Dalvaux. Quelques confrères ou consoeurs veulent-ils prendre Ποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, Νομίζω ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Τερβό για την καλή εργασία που έκανε και νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακριβώ, όπω τα λέει. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα για να καταστούν οι ζωέ των ανθρώπων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πιο απλά σε ό,τι αφορά τα δημόσια έγγραφα. Συμφωνούμε λοιπόν με την ιδέα τη διαβρύνση παιδιαφαρμογής. Συμφωνούμε με την υποχρέωση πληροφόρηση των πολιτών από πλευρά των πρώτων μελών για την κατάσταση που ισχύει. Νομίζω λοιπόν ότι την Πέμπτη θα γίνει η τριμερή διάλογο. Ελπίζουμε να αποκομίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με την εργασία που έκανε η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κυρία Ρόταλα. Άλλοι συνάδελφοι θα ήθελαν το λόγο. Όχι. Αν μου επιτρέπετε να κάνω εγώ δύο προσωπικές παρατηρήσεις για αυτό το θέμα τις είχα ήδη προετοιμάσει χωρίς να πιστεύω ότι, χωρίς να ξέρω τι θα προεδρεύσω εν πάση περιπτώσει πρώτον στις προτάσεις του Συμβουλίου ε, χρησιμοποιείται η λέξη notary public η οποία αντικαταστάθηκε από τη λέξη notary νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τη διάκριση ανάμεσα στις δύο διαφορετικές αυτές πράξεις και να διατηρήσουμε την έκφραση Notary Public. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε κυρία Ντελβό. Οπότε δεν θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Ε, οι solicitors, αυτοί του Βρετανοί, του οποίου αποκαλούμε solicitors, επικυρώνουν μόνο την υπογραφή, όχι το περιεχόμενο του εγγράφου. και εμείς ε, κάνουμε τέτοιου είδους διακρίσεις. Μπορούμε ε, να έχουμε ε, μια επικύρωση του γνησίου της υπογραφής που είναι ένα πράγμα και άλλο πράγμα είναι ο έλεγχος του περιεχομένου. Μετά, η προτρόταση τροπολογίας μάλλον οι προτάσει μα βρίσκουν σύμφωνο νομίζω για την τροπολογία 6 στο άρθρο 5 όμω, παράγραφο παράγραφος 1α ε, έχω το εξή σχόλιο ο κανονισμός δεν θα πρέπει να επιτρέψει οποιαδήποτε απάτη. Όμως, αν δεχτούμε, αν δεχόμαστε ε, μη επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δημιουργηθούν παράθυρα για απάτες και να αρχίσουν να κυκλοφορούν, να αρχίσουν να κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός ε, πλαστών εγγράφων, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναδείτε αν θέλετε αυτή την τροπολογία. Κομισιόν, θα ήθελε το λόγο. Où est-elle Oui. Non Όχι. Η κυρία Βίλα είναι εδώ, θέλει να πάρει το λόγο. Η Κομισιόν δεν θέλει να πάρει το λόγο. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελπό. Ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες σας, κύριε Τελβό. Η Λεξιβουριανή Προεδρία θα ήθελε να κλείσει το θέμα πριν το τέλος του εξαμήνου. Και εμείς επιθυμούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Έχει, έχουμε ήδη καθυστερήσει. Οπότε ελπίζω ότι ο τριμμένος διάλογος θα πάρει μερικές συναντήσεις, λίγες, έτσι ώστε να κλείσει το θέμα. Ελπίζω σε κανένα μήνα να έχουμε καταλήξει. Ωραία. Ελπίζω. Δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Ευχαριστούμε. Ε, επαναλαμβάνω ότι περιμένουμε το όνομα του συναδέλφου που θα αντικαταστήσει τον κύριο Μάριο. Περι... Α, θα είναι ο κύριος Παβέλ Τέλιτσκα. Ωραία, εντάξει, ενημερωθήκαμε και γι' αυτό. Περνάμε στην επόμενη, στο επόμενο θέμα. Έκθεση Χαουτάλα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πρόταση για γνωμοδότηση της Γιούρη, για μία αναθεώρηση μιας πρότασης κανονισμού που προστατεύει κατά των επιπτώσεων της ε, εξοεδαφικής εφαρμογής της νομοθεσίας που υιοθετείται από μια τρίτη χώρα και των δράσεων που βασίζονται πάνω σε αυτήν ή απορρέουν από αυτήν. Ο στόχος του κανονισμού είναι να προστατεύσει τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων εναντίον οποιονδήποτε επιπτώσεων της εξοδαφικής εφαρμογής της νομοθεσίας. Τα τα νομοθετήματα αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού και συμπεριλαμβάνουν τις κυρώσεις του 96 του Ιράν και της Συρίας και η πράξη της αλληλεγγύης ε, για την Κούβα του 96 των Πολιτειών και την προστασία ή κίνηση των κεφαλαίων που αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες κοινότητας και τρίτων χωρών. Εάν ένα δικαστήριο ή παρόμοια αρχή αποφασίσει κατά των οικονομικών ή χρηματοπιστωτικών συμφερόντων ενό φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να βασίζεται σε νομοθετήματα που αναφέρονται σε αυτό το παράρτημα, η απόφαση αυτή δεν θα αναγνωρίζεται ή δεν θα είναι εκτελεστή. Ε, Συν το χρόνο, αυτό ο κανονισμό έχει τροποποιηθεί πλήστε φορέ. Η Κομισιόν τώρα θέλει να κάνει μια κωδικοποίηση και αυτή η κωδικοποίηση σκοπό να καταστήσει τον κανονισμό ακόμα μια φορά σαφή και διαφανή. Η Κομισιόν θα ήθελε να κάνει και κάποιες ουσιαστικέ αλλαγές και αυτή η πρόταση παρουσιάζεται υπό τη μορφή μιας αναθεώρησης, recast. Για να μπορέσει η Επιτροπή μας, η Γιούρη, να κάνει μια γνωμοδότηση, ε, μια γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας των τριών νομικών υπηρεσιών, του Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και του Συμβουλίου, απαιτείται με βάση το άρθρο 103 και τη διαθεσμική συμφωνία για τις αναθεωρήσεις εν γέννη. Για να υπάρξει γνωμοδότηση για το αν η πρόταση αποτελεί απλή κωδικοποίηση χωρίς καμία αλλαγή της, της ουσίας και επειδή δεν έχει εκδοθεί ποτέ τέτοια γνωμοδότηση, αυτή τη στιγμή όμως αυτή η γνωμοδότηση εκδοθεί, τότε η Επιτροπή Γιούρη θα πρέπει ε, να γνωμοδοτήσει αφού εκδοθεί η, Επιτροπή, η γνωμοδότηση δηλαδή, της Επιτροπής αυτής των τριών νομικών υπηρεσιών. Θα ήθελα λοιπόν τώρα οι τρεις νομικές υπηρεσίες να μας ενημερώσουν για την γνωμοδότηση που υποτίθεται ότι εμείς θα πρέπει να ετοιμάσουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Τελειώσατε την παρουσίασή σας. Πολύ ωραία. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Μεντόλα. Που εκπροσωπεί την νομική υπηρεσία. Thank Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση αναθεώρησης, συναντηθήκαμε δύο φορές με την Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας των Τριών Νομικών Υπηρεσιών, αλλά δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε μέχρι στιγμής. Το βασικό πρόβλημα αφορά την πιστοποίηση, το πιστοποιητικό που θα πρέπει να εκδώσει η συμβουλευτική ομάδα για τη χρήση της διαδικασίας κωδικοποίησης επί της πρότασης. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η πρόταση που αναθεωρούμε βασιζόταν σε τρεις νομικές πράξεις του εντάξει εμπορική πολιτική, ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και τη λεγόμενη ρήτρα ευελιξίας. Τώρα, επ' ευκαιρία της αναθεώρησης, φαίνεται ότι η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου θεωρεί ότι για να βελτιώσουμε την πρόταση, η ρήτρα ευελιξίας το άρθρο δηλαδή 352 της συνθήκης αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να απαλληφθεί από την πρόταση. Ενώ οι άλλες νομικές υπηρεσίες της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου δεν συμφωνούν με αυτό το συμπέρασμα. Όχι γιατί δεν είμαστε υπέρ της απαλληφής, της ρήτρας ευελιξίας, αλλά γιατί θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή καθεαυτή απεικονίζει το κείμενο όπως είχε δημιουργηθεί το 1996 μετά από δύο συναντήσεις λοιπόν, γι' αυτό έχουμε φτάσει αδιέξοδο. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ουδής. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 6 της Μεσίας Διάταξης. Η κυρία Ζωέλ Μπερζερόν έχει το λόγο. Η κυρία Μπερζερόν, παρακαλώ. Κυρία Μπερζερόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η προστασία των ευάλωτων ατόμων είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Δυστυχώς, όλοι μας είμαστε ενδυνάμει ε, ευπαθείς ενήλικες. Κάποια στιγμή, ας πούμε, θα το αντιμετωπίσουμε ή κάποιος οικείος. Εξαιτία της παράτασης του προσδόκιμου ζωής, τα άτομα που είναι πάνω από 80 χρονών είναι 50 εκατομμύρια στην Ευρώπη και με βάση την ΕΟΚΕ θα είναι 137 εκατομμύρια το 2025. Η εξάρτηση, η ψυχική και ψυχολογική υγεία, όπως ε, το Αλτχάιμερ, ε, ή και άλλες ψυχοπαθολογίες μας αναγκάζουν να αγγίψουμε από του προβλήματος. Οι ευπαθείς ενήλικες δεν είναι μόνο άτομα ηλικιωμένα, αλλά όλα τα άτομα των οποίων οι φυσικές ή πνευματικές ικανότητες είναι μειωμένε. Στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μια αφύπνιση οδήγησε σε μια αναθεώρηση των διαφόρων συστημάτων. Στη Γαλλία το 2007 ε, δημιουργήθηκαν διάφοροι βαθμοί εξάρτησης από την ε, προστασία έως την πλήρη ανάληψη. Και οι κυδεμόνες αυτοί ε, διαχειρίζονται αυτά τα ευπαθή άτομα. Ποιοι είναι αυτοί οι ευπαθείς ενήλικες. Είναι ενήλικες, έτσι, και δεν είναι ανήλικοι. Είναι άτομα φυσικά, τα οποία είναι πάνω από 18 χρονών, που είναι η ηλικία ενηλικίωση στην Ευρώπη, εκτός από την ε, Σκοτία που η ηλικία αυτή είναι στα 16 χρόνια. Είναι ε, προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση ανικανότητα να διαχειριστούν και το άτομό τους αλλά και τα αγαθά τους και θα πρέπει να τους ε, συνοδεύουμε. Ε, στην Ευρώπη έχουμε την ε, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στον ευρωπαϊκό χώρο τα προστατευόμενα άτομα ή τα ενδυνάμει προστατευόμενα θα πρέπει, ε, μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν σε διάφορες χώρες της Ένωση. Ένα παράδειγμα, ένας ε, ε από τις σκανδιναβικέ χώρες θέλει να περάσει ας πούμε ε, τη ζωή του μετά τη σύνταξη σε μια, πιο, μια χώρα ας πούμε με πιο ήπιο χρήμα που δεν είναι ε, η χώρα του ε, οι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν στη χώρα τους μετά από χρόνια που έχουν ζήσει στο εξωτερικό. Ε, επίσης, ε, είτε γιατί παντρεύεται κανείς, είτε ε, κάνει κανείς συνάπτει ένα γάμο ας πούμε, με ένα ξένο, άλλο υπήκο, υπήκο άλλου κράτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γιατί για επαγγελματικού λόγους θέλει να ταξιδέψει. Ε, το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε την περιουσία του όταν τα άτομα αυτά, την περιουσία του όταν τα άτομα αυτά θα δυνατούν να το κάνουν. Ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ειδικέ νομοθεσίες, αλλά δεν υπάρχει νομική ομοιομορφία. Μία συγκριτική μελέτη των διαφόρων καθεστώτων προστασίας των ανίκανων ε, ενηλίκων έγινε το 2008 από το Ελβετικό Ινστιτούτο ε, του Συγκριτικού Δικαίου της Λοζάνης για τη Γερμανία, για την Τσεχία, την Μεγάλη Βρετανία, την Ρουμανία και τη Σουηδία και τη Γαλλία. Και έδειξε πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών των χωρών αυτή η μελέτη του Ινστιτούτου να σας δώσω τα ισχύοντα κείμενα, διεθνή κείμενα, τα οποία προς το παρόν διέπουν ε, τα άτομα αυτά. Ε, το, τα πιο σημαντικά, έτσι. Είναι η Σύμβαση της Χάγης της 13ης ε, Ιανουαρίου 2000. Καθορίζει τα ενήλικα άτομα που είναι ευπαθή και λέει ότι είναι ενήλικες που λόγω μιας α, μείωσης των προσωπικών τους ικανοτήτων δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό το κείμενο ε, αφορά τα υλικά συμφέροντα του ενηλίκου, αλλά και το σεβασμό του, την ε, ζωή του και την αξιοπρέπειά του. Ε, υπάρχει μια ευρεία έννοια του, της, του ευάλωτου και αφορά και τους με, πρόσφυγες ή μετακινούμενους. Ανάλογα το κράτος της συνήθους κατοικίας είναι υπεύθυνες ε, οι αρμόδιε αρχέ. Η Σύμβαση της Χάγη είναι ένα καλός σύνολο κανόνων, σαφών, ε, συνεκτικών, ε, κατάλληλο για τον μοντέρνο κόσμο και η επαφή με τον διαφόρων αρχών είναι βασικό στοιχείο της Σύμβασης. Αυτό το κείμενο αφορά την προστασία των ατόμων που μας αφορούν και είναι το πιο ε, βελτιωμένο σε ό,τι αφορά το διεθνές δημόσιο δίκαιο. Ε, μόνο δυστυχώ όμω 14 άτομα το έχουν υπογράψει. Μπορεί να κάνω λάθο, αλλά νομίζω 6 χρόνια το επικύρωσαν κιόλα, το οποίο είναι εντελώ ανεπαρκέ για να εξασφαλίσουμε την ε, εφαρμογή του. Ε, για να μπορεί να αδύνατον. Μπορούμε να αναφέρουμε τη σύμβαση του ΟΗΕ τη 13η Δεκεμβρίου του 2006 που μπήκε το Μάιο του 2008 και που αφορά τα ανάπηρα άτομα. Ενισχύει τι υποχρεώσει ό,τι αφορά τις, την αναγνώριση νομική προσωπικότητας του άτομου σε συνθήκες ε, ισότητα και διεθνούς συνεργασίας. Άλλο διεθνές μέσο είναι η σύσταση του 23 Φεβρουαρίου του 1989 της Επιτροπής ε, Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφορά την προστασία των ανίκανων ε, ενηλίκων και μιλάει για τις αρχές που διέπουν την βοήθεια και την εκπροσώπηση των ευπαθών ενηλίκων σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν ε, την προσωπικότητά του ή τα αγαθά του. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ευθύσει την προσοχή τη Κομισιόν στην ε, ανάγκη να νομοθετήσει σε ό,τι αφορά την προστασία των ατόμων αυτών. Μία έκθεση πρωτοβουλία είχε δοθεί σε έναν συνάδελφο, τον κύριο Αντώνιο Λόπε Ιτούρε. Ε, η έκθεση αυτή μιλάει για την ανάγκη προστασία νομική διασυνοριακού χαρακτήρα και μιλά για τη ουσιαστική σημασία της ε, σύμβασης της Χάγης και έδινε κίνητρα για την επικύρωση των ε, υπογραφωμένων. Έδινε τη δυνατότητα σε δύο κράτη-μέλη επίσης να προσαρτήσουν σε αυτή την ε, σύμβαση απλώς και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ. Υπάρχουν πέντε, ε, πέντε σημεία ε, για τους, τις βασικές αρχές της πρότασης αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. White. Να προωθήσουμε την αναγνώριση και εκτέλεση των νομικών αποφάσεων ή διοικητικών αποφάσεων που αφορούν τα άτομα τα οποία ε, χρήζουν προστασία. Να δημιουργήσουμε διατάξεις για να υλοποιήσουμε τους στόχους, να υπάρχει ένας χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, διευκολύνοντας την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων, ε, τα οποία θέλουν, ε, σκοπό έχουν την προστασία. Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών επίση, για να εφαρμοστεί ο νόμο. Να δημιουργούν ειδικά μέτρα για τη συνεργασία των κρατών μελών, βασιζόμενοι στα εργαλεία τη ε, Σύμβαση τη Χάγη. Να δημιουργηθεί. Κοινά, ε, να δημιουργηθούν κοινά έντυπα για να υπάρξει η ενημέρωση για τι αποφάσει προστασία και να κυκλοφορούν ε, οι αναγνωρίσεις και εκτελέσεις των πράξεων. Να δημιουργήσουμε ένα νέο ε, κοινοτικό έντυπο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εντολή ανικανότητας και που θα ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρότι η έκθεση αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της Νομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου και μερικά εξακολουθούν να εδρεύουν εδώ, δεν υπήρξε συνέχεια από πλευρά Κομισιόν. Και ακριβώ για αυτό το λόγο παίρνουμε την πρωτοβουλία σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Προτείνουμε να αποτελέσει ε, βάση εργασία αυτέ οι αρχέ. Ο χώρο δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα που επιτρέπουν στα ευπαθή άτομα να κυκλοφορούν ελεύθερα στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προστατεύονται από διοικητικά ή νομικά μέτρα που αναγνωρίζονται από όλους. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η δικαστική συνεργασία ε, για τι αστικέ υποθέσει μεταξύ των κρατών μελών, άρθρα 65 και 61 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημιουργία κοινών ε, ευρωπαϊκών εντύπων ε, για την διάχυση τη πληροφορία των μέτρων προστασία, χωρί να ξεχάσουμε και το σεβασμό, τη θέληση και την αυτονομία των ατόμων αυτών. Συμπερασματικά. Ποιο είναι το συμφέρον ενός ευρωπαϊκού κειμένου, ποιο είναι το νόημα. Η σύμβαση της Χάγης για τα άτομα αυτά είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει επικυρωθεί μόνο από έξι χώρε. Δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσουμε το πρόβλημα των ευπαθών ατόμων αυτών διασυνοριακά στην Ευρώπη. Η απουσία μια δεσμευτική ρύθμιση για τα κράτη-μέλη ε, ζημιώνει την προστασία ε, των ατόμων αυτών και το κόστο είναι 16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όπω εκτιμάται. Λόγω τις ανάγκες να ξεκινήσει εκ νέου διαδικασία εφαρμογής μέτρων προστασίας ανάλογα με τη χώρα που μετακινείται το άτομο, αλλά και γιατί υπάρχουν και ζημίες για τα συμφέροντα, τα οικονομικά των ατόμων αυτών που δεν προστατεύονται επαρκώ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κανονισμό, ο οποίος θα βασίζεται στη βελτίωση, εάν είναι δυνατόν, ε, τη σύμβαση της ε, καλύτερα κανονισμός παρά οδηγία, γιατί ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ε, ημερομία που αναφέρει ή το πολύ πολύ 20 μέρες μετά, μετά τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν επιλεκτικά ημερικώ. και δεν χρειάζεται μια εθνική μεταγραφή για να τεθεί σε ισχύ. Αντίθετα με την οδηγία, το που γίνεται δεσμευτική, μόνο όταν έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ε, Κομισιόν, μπορώ να σας ρωτήσω γιατί δεν δόθηκε καμία συνέχεια το κείμενο αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2008, στην έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου White. Υπήρξε και ένα ερωτηματολόγιο του 2014 που απευθύνεται στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της Σύμβασης της Χάγης και τίποτα άλλο. Ποιε είναι οι δυσκολίε οι ιδιαίτερες που εντόπισε η Κομισιόν που συνδέονται με αυτή την εφαρμογή τη σύμβαση αυτή. και τι συνέχεια θα δώσετε στη δική μα έκθεση πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Merci à vous. Euh. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Με διευκολύνεται να δώσω το λόγο στην κυρία Πατρίσια Ντελούκα από την Κομισιόν ε, για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Um, Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς από πλευράς μας ο συνάδελφος δεν έχει καταφέσει ακόμα μπορούμε να σας απαντήσουμε γραπτά, αν θέλετε, πολύ λυπούμαστε, ή όπως επιθυμείτε, μας περιπτώσει. Ε, καταλαβαίνω το μέγεθος της θλίψης σας. Ε. ε, θέλει κανένα άλλο μέλος να πάρει το λόγο. Κυρία Κομοντίνη. Thank um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω και από το ΕΛΚ για την έκθεση αυτή, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίασή τη και που μας παρουσίασε και τα πιο βασικά ζητήματα τα οποία είχαμε εντοπίσει και στην προηγούμενη εργασία μας από πλευρά του Κοινοβουλίου. Πώς βλέπουμε στην έκθεση. Γιατί νομίζω ότι όλοι εδώ Θέλουμε να προστατεύσουμε τα ευάλωτα αυτά άτομα. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία επ' αυτού. Είναι πολύ ατυχέ που πολλά κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν επικυρώσει τη συνθήκη τη Χάγη. Και προσπαθούμε να αναζητήσουμε έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε τα ευάλωτα άτομα σε διασυνοριακές καταστάσει. Άρα, προσβλέπω να ακούσω προτάσεις ε, για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, όπως η αναγνώριση ενάμικων διαδικασιών, όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών, ε, διαφορές ε, επίσης μεταξύ των συμβολιογραφικών πράξεων, τα οποία, οι οποίε χρησιμοποιούνται για από τα ευάλωτα άτομα σε ό,τι αφορά και τα περιουσιακά στοιχεία σαν διασυνοριακέ συναλλαγέ. Ωστόσο, θα ήθελα και εγώ να ακούσω την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση που θέσατε. σε ό,τι αφορά κυρίως την έλλειψη αντίδρασης στις προτάσεις που έχει κάνει στο παρελθόν το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, άλλοι συνάδελφοι. Ωραία, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απευθύνω ε, μια, ένα αίτημα προς την Κομισιόν. Είναι ένα θέμα που χρονίζει. Γι' αυτό λόγο απάντηση θα θέλαμε να μας δοθεί αυτό το μήνα. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Θα μεταφέρω το αίτημά σας στην αρμόδια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ποιο είναι το όνομα και η θέση της υπεύθυνης του υπεύθυνου για αυτό το θέμα στην Κομισιόν. Uh, ε, ενημερώθηκε ε, ο συνάδελφος και δεν κατάφερε να έρθει ε, για λόγους που δεν γνωρίζω, λυπάμαι, δεν είναι παρούσα. Σημειώνω όμως το ερώτημά σας και θα σας απαντήσουμε γραπτός ή δυνατόν μέχρι το τέλος του μήνα όπως ζητήσατε. Οπότε αυτό το, αυτό το άτομο δεν έχει όνομα. Ε, already... Το είπατε το όνομά σας. Το όνομα της ε, στην αρχή. Εσείς το, το αναφέρατε. Α, ah, πρόεδρος. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο και δεν έχει αλλάξει. Ωραία. Παρακαλώ πολύ ενημερώστε την ότι αναμένουμε με ανυπομονησία την απάντησή τη. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησίας διάταξη. Ε, έκθεση του κυρίου Ράντεφ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εδώ και αρκετό καιρό περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις για κοινά ελάχιστα πρότυπα πολιτικής οικονομίας. Και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία να εργαστεί για αυτό το θέμα και ορίστηκα εισηγητής. Η ελεύθερη κυκλοφορία δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνθηκε μετά την κατάρριξη του Σεκουάτουρ και αυτό κατέστη πιο, κατέστησε πιο, ε, πιο εύκολη την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων. Αλλά α, για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ε, μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να τηρούνται κοινοί οικονομικοί κανόνε. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι κάτι περίπλοκο και είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αφενός έχουμε τα ήπια μέσα όπως την κατάρτιση, επιμόρφωση των δικαστικών, ανταλλαγές καλών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δικαστών κλπ. κλπ. Απ' την άλλη μεριά η αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, σημαίνει επίσης ότι θα, ε, τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν τους ίδιους κανόνες πολιτικής δικονομίας. Η νομοθετική παρέμβαση για κοινά ελάχιστα πρότυπα πολιτική οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει ε, ε, ένα τρόπο για να εδραιωθεί η αμοιβή εμπιστοσύνη. Και έχουμε μέσα που μπορούν να μας βοηθήσουν μέσα σε εθνικό επίπεδο αλλά ε, και εννοώντας ε, την ε, διαδικασία ανάκτησης ε, μικρών χρεών, την επιγραμμική επίλυση διαφορών και διάφορα άλλα μέσα. Έχουμε επίσης και οδηγίες, τομεακές οδηγίες, όπως για παράδειγμα στον τομέα του προστασίας του καταναλωτή, της ομαδικής ιδιοκτησίας και του δικαίου του ανταγωνισμού. Αυτές ε, είναι οδηγίες οι οποίες δεν άπτονται την πολιτική, της πολιτικής οικονομίας στο σύνολό της, αλλά ορισμένων πτυχών της μόλων. Για παράδειγμα, ε, η οδηγία ε, δωρεάν νομικής υποστήριξης ενώ εμείς την πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εναρμονίσουμε την κανόνες πολιτικής δικονομίας. Τέτοιου τύπου εναρμονίσεις βέβαια είναι προβληματικό, προβληματικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ε, χρειαζόμαστε όμως μια οριζόντια οδηγία η οποία θα οδηγούσε σε σύγκληση τα εθνικά νομικά συστήματα των κρατών μελών. Έτσι θα αυξανόταν η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα ε, συστήματα των κρατών μελών και θα εγγυόμασταν έτσι ε, ε την απονομή της δικαιοσύνης. Το Μέο του 2014 ξεκίνησε το πρώτο βήμα, το Ευρωπαϊκό Νομικό Ινστιτούτο συναντήθηκε με το Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου και ξεκίνησαν μια κοινή πρωτοβουλία με στόχο να διαπιστωθεί αν οι αρχές της UNIDROA και οι αρχές του Αμερικανικού Ινστιτούτου θα μπορούσαν να ε, προσαρμοστούν στην ευρωπαϊκή κατάσταση. Στις αρχές του 2015 οι πρώτες, τα πρώτα πορίσματα ε, παρουσιάστηκαν τα πρώτα πορίσματα και δημιουργήθηκαν καινούριε ομάδες εργασία. Τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή μας με τους ε, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ε, Νομοθεσίας ε, πτυχές αυτών των προβλημάτων. Και έχουμε πολλά προβλήματα, πολλά και διάφορα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις εθνικές δικονομ... αρχές πολιτικής οικονομίας. Και χρειαζόμαστε ένα κείμενο που θα βελτιώσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη Θα πρέπει οι καινούργιοι κανόνες να ε, διευκολύνουν και όχι να περιπλέκουν την κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι ο βασικός στόχος μας είναι να εργαστούμε προς το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να ε, χαίρουν των ίδιων οικονομικών δικαιωμάτων. Και στο διοικητικό δίκαιο και στο ποινικό δίκαιο. Όχι μόνο στο αστικό δίκαιο. Όμως ακούω ότι οι ειδικοί θα καταφέρουν να βρουν μια λύση έτσι ώστε ε, να επιτρέψουν στην Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις. Ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλιά σας και αυτά της Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε κύριε Ραντεύ. Και θα ζητήσουμε τώρα να μας πει δυο λόγια η Κομισιόν αν επιθυμεί. Και συνεχεία θα ακούσουμε τους συναδέλφους εάν θέλουν να πάρουν το λόγο. Η Κομισιόν θέλει να μιλήσει για το, την έκθεση ράντεβ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ. Νόρα Ρόσνερ ονομάζομαι και είμαι από την DG Justice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ανταλλαγή αυτή απόψεων που διοργανώθηκε για το θέμα αυτό το πολύ σημαντικό. ορίζουμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα κοινά ελάχιστα πρότυπα πολιτική δικονομία και θεωρούμε ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν ε, πολύ μεγάλη σημασία και σε ποινικέ αλλά και σε αστικέ υποθέσει. Και όντω, ε, όταν υπάρχει άρνηση αναγνώριση τέτοιων αποφάσεων, ε, αυτό οφείλεται στην. Στις διαφορές που υπάρχουν στην πολιτική δικονομία. Ο σεβασμό λοιπόν των δικαιωμάτων αυτών των μερών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο πάνω στο οποίο βασίζεται η εύρυθμη λειτουργία των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει από τους δικαστές και από τους ε, νομικούς απόλυτη εμπιστοσύνη σε αποφάσεις άλλων ε, κρατομελών. Αυτό κοινοποιήθηκε στην στο σχετικό έγγραφο για τη δικαιοσύνη 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ληφθούν υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία και να διασφαλίζονται πάντα τα, συμφέροντα των παιδιών σε τέτοιε νομικέ διαδικασίε. Εκ παραλίλου, τέτοια εργαλεία σε διαφορετικό βαθμό περιλαμβάνουν και κανόνε πολιτική οικονομία. Οικονομικού κανόνε. Οι ευρωπαϊκέ διαδικασίε, ε, όπω αναφέρει ο εισηγητής, ε, μικρές αξιώσεις χαμηλών ποσών για την πληρωμή μικρών ποσών, αλλά και άλλοι δικονομικοί κανόνες που περιλαμβάνονται σε άλλα ε, όργανα, σε άλλα εργαλεία όπως ο κανονισμός σε 1 και Βρυξέλλες 2. Επιπρόσθετα, τα πρότυπα που ορίζονται σε διάφορα μέσα πολιτικές οικονομίες Υπάρχουν διάφορα πρότυπα τα οποία έχουν επιβληθεί από το δικαστήριο για να εξασφαλιστεί η σωστή προστασία των πολιτών και να είναι αποτελεσματικοί οι κανόνες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει δράση σε ό,τι αφορά την πολιτική οικονομία. Κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση της, ε, των ε, εγγράφων και της ε, χρήση τους στα κρατη για να δούμε πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός και για να βρεθούν τομείς που ενδεχομένως ε, ε, ζητούν δράση ε, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω για παράδειγμα η διασυνοριακή επίδοση γράφων. Θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον αυτό αποτελεί μια δυνατότητα, λαμβάνοντα υπόψη και την δυνατότητα των μερών και την μείωση του οικονομικού κόστου. Επίσης θα ξεκινήσει αξιολόγηση των εθνικών πρακτικών και νόμων σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της ελεύθερης ε, μεταφοράς των δικαστικών αποφάσεων. Τέλος. Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να προσθέσω ότι η πρωτοβουλία, όπως η ανταλλαγή αυτή απόψεων που οργανώνεται σήμερα, είναι γεγονότα που τα καλωσορίζουμε είναι επωφελή στοιχεία για την όλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέρη τα οποία θα δίδουν πληροφορίες. Ε, αυτό είναι ένας πρακτικός τρόπος για να εργαστεί κανείς. Οι συνάδελφοί μου θέλουν να πάρουν το λόγο. Ουδής. Ουδής. Η κυρία Χάουταλα. Σας ευχαριστώ. Μια ερώτηση μόνο να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς τον εισηγητή. Ποια είναι τα διδάγματα από την επιτυχία των ελάχιστων ε, κανόνων για τις ε, ποινικέ διαδικασίες. Φυσικά υπάρχουν διαφορές και είναι σημαντικές, αλλά υπάρχουν ε, οποιαδήποτε μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τη σύγκριση αυτή. D'abord, si vous voulez. Κύριε Ράντεφ, αν θέλει να απαντήσει την κυρία Χάρτελα. Ευχαριστώ. Όταν υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα, μειώνεται η ασάφεια. Το βλέπουμε αυτό στο ποινικό δίκαιο και στη, στον κώδικα ποινική δικαιοδικονομίας. Και έτσι αρχίζει να λειτουργεί καλά η δικαιοσύνη προ το συμφέρον των πολιτών. Εδώ μιλάμε για τα συμφέροντα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί ο καθένας έχει διάφορες αστικές σχέσεις Όταν αρχίζουμε να κωδικοποιούμε τα πρότυπα, νομίζω ότι αυτό ε, μόνο ωφέλη μπορεί να δώσει. Και αυτά τα ωφέλη θα αφορούν, θα συμπεριλαμβάνουν και αύξηση της ε, εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και απλέ, απλούστερες διαδικασίες για τους πολίτες. Η Κομισιόν θέλει να απαντήσει την κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, πολιτικής δικονομίας είναι το δικαίωμα των διαδίκων, των μερών, πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκη δίκη. Και εδώ υπάρχουν κάποιες ομοιομορφίες με το ποινικό δίκαιο. Αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο. Δηλαδή, στο αστικό δίκαιο έχουμε διασυνοριακή αναγνώριση και εφαρμογή των αποφάσεων στην Ευρώπη. Ενώ στο ποινικό δίκαιο τα πράγματα είναι κατά τη διαφορετικά. Κανοποιηθήκατε κυρία Χάουτελα. ή θέλετε να κάνετε δευτερεύουσες ερωτήσεις. Όχι. Μια και είμαστε αρκετά μπροστά. Έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα δηλαδή. Θα ήθελα να επανέλθουμε λιγάκι στην έκθεση της κυρίας Μπεοζερό, γιατί το άτομο προς το οποίο απευθύνατε τις ερωτήσεις σας, η κυρία Ντελούκα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι παρούσα. Κυρία Μπεοζερό, θα μπορούσατε να ξαναρωτήσετε τα ίδια πράγματα στην κυρία Ντελούκα και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε και διάλογο οι δυο σας. Ρωτούσα την Κομισιόν γιατί δεν έχει δοθεί καμία συνέχεια στην έκθεση πρωτοβουλία του κυρίου White το 2008 απλώς ένα ερωτηματολόγιο είχε απευθυνθεί το 2014 στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή τη σύμβαση τη Χάγη, που είναι ουσιαστική για την αντιμετώπιση των ευπαθών ενηλίκων. Ποιε είναι οι δυσκολίε που εντόπισε η Κομισιόν και που εμπόδισαν το να δοθεί συνέχεια στην έκθεση πρωτοβουλία και να εκπνεύσει και τι συνέχεια σκοπεύετε να δώσετε στην έκθεση πρωτοβουλία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Προέκυψε ένα μικρό πρόβλημα. Να απαντήσω όμως την πρώτη σας ερώτηση. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν δόθηκε καμία συνέχεια στο ψήφισμα του 2008. Να σας θυμίσω ότι το ψήφισμα του 2008, στην πρώτη του παράγραφο, ζητούσε από την Κομισιόν ε, μόλις ε, αποκτηθεί επαρκής εμπειρία από την εφαρμογή της σύμβασης να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια νομοθετική πρόταση. Ο όρος ήταν λοιπόν να έχουμε αποκτήσει αρκετή πείρα από την εφαρμογή της σύμβασης. Η σύμβαση, όπως γνωρίζετε, ετέθησε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2009. Το 2008 ήδη η Κομισιόν είχε ζητήσει από τα κράτη-μέλη και τους είχε, τα είχε ενθαρρύνει να επικυρώσουν τη σύμβαση. Στην σύμβαση δεν υπάρχει ρήτρα που να επιτρέπει την επικύρωση συνθήκη από διεθνείς οργανώσεις ή διεθνείς οργανισμούς όπως η διεθνει οργανισμου οπως Ένωση. Μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να την επικυρώσουν. Ε, οργανώσαμε μια πρώτη συζήτηση στο Συμβούλιο το 2010. Η Κομισιόν ζήτησε αυτή τη συζήτηση προκειμένου να καταγράψουμε την κατάσταση. Αρκετά κράτη-μέλη απάντησαν στο ερωτηματολόγιο λέγοντας ότι βρίσκονται στην διαδικασία εξέτασης της σύμβασης ε, εν ώψη επικύρωσής της. Καθώς δεδομένου ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης προέβλεπε ε, μια παρακολούθηση από την Κομισιόν του 2014, οργανώσαμε μια δεύτερη συζήτηση αυτού του θέματος με ένα πιο λεπτομερές ερωτηματολόγιο που απευθύναμε στα κράτη-μέλη προκειμένου να μας ενημερώσουν για το ποιες είναι οι δυσκολίες και γιατί δεν έχουν ακόμα επικυρώσει τη σύμβαση. Μέχρι σήμερα μόνο 7 κράτη-μέλη την έχουν επικυρώσει. Το πρώτο, α, τα πρώτα αποτελέσματα ήταν εθαρρυντικά μπορώ να πω γιατί πολλά κράτη-μέλη αρκετά ανέφεραν ότι βρίσκονται στο τέλος της εσωτερικής τους διαδικασίας που οδηγεί στην επικύρωση. Για παράδειγμα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία. Και ένας άλλος σημαντικός αριθμός κρατών μελών είπαν ότι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση επικύρωσης της σύμβασης και προσχώρησης αυτήν. Δεν υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην ίδια την επικύρωση. Δύο προβλήματα μας υπογραμμίστηκαν από τα κράτη-μέλη κυρίως. Πρώτον, ότι δεν είναι και πολλές οι περιπτώσεις προστασίας ευάλωτων ενηλίκων. Οπότε δεν βλέπουν την ανάγκη μιας νομοθετικής πράξης για την επικύρωση αυτής της σύμβασης. Και η άλλη δυσκολία είναι το κόστος. Γιατί φοβούνται κάποια ότι το σύστημα ε, που προβλέπει τον καθορισμό κεντρικών αρχών κλπ. θα δημιουργούσε πρόσθετα κόστη. Αυτές είναι οι δύο δυσκολίες τις οποίες μας ανέφεραν. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Θα επανεξετάσουμε μαζί με τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερος με αυτά που είπαν ότι βρίσκονται κοντά στην επικύρωση θα τους ξαναρωτήσουμε για ποιο λόγο δεν έχουν επικυρώσει ακόμα τη σύμβαση ε, και ενώ θα καταγράψουμε ταυτόχρονα και την κατάσταση σε ό,τι αφορά τα άλλα κρατημέλη που αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει ομάδες εργασίας και εξετάζουν τη σύμβαση. Λίγα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία δεν σκοπεύουν οριστικά να την επικυρώσουν. Τώρα, για τα κράτη τα οποία έχουν ήδη επικυρώσει τη σύμβαση, ε, θα τους ε, ρωτήσουμε, θα τα ρωτήσουμε ποια είναι η εμπειρία τους, αν Μάλλον τα ρωτήσαμε ποια είναι τα προβλήματα που προέκυψαν, ποια είναι η εμπειρία τους. Μας απάντησαν ότι είναι καλή η σύμβαση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν και πολύ πρακτική εμπειρία γιατί οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες. Ευχαριστώ. Madame Bergeron, vous avez reçu satisfaction. κυρία Bergeron τουλάχιστον απάντηση πήρατε. Καταπλήσωμε, εκπλήσωμε που, υπάρχουν, που λένε τα κράτη-μέλη ε, λένε ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διάφοροι συνταξιούχοι φεύγουν. Εγώ νομίζω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια ο άνθρωπος ε, δικαπλασιάστηκαν τα άτομα αυτά. Ε, σε ένα χωριό, εν είχαμε 6.000 ανθρώπου και έχουμε τώρα χιλιάδες. Πολλές χιλιάδες. No, no, ναι. Συμφωνώ με την κυρία Ζερόν. Όλο και περισσότερε περιπτώσει εμφανίζονται, Ορισμένε ε, κοινοποιούνται στην Κομισιόν, άλλες όχι. Αλλά κάποια κράτη-μέλη προφανώς δεν έχουν και πολλή εμπειρία ακόμα. Χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλιο και η Γερμανία έχουν κάποιες περιπτώσεις. Άλλα κράτη-μέλη είπαν ότι ποτέ δεν αντιμετώπισαν τέτοιες περιπτώσεις. Και σας θυμίζω ότι πρόκειται για τις διαμεσοριακές ε, περιπτώσεις, έτσι. Όχι για την ε, προστασία ε, χώρας το εσωτερικό της χώρας, στην επικρατεία της. Μιλάμε για διασυνοριακές ε, ε, υποθέσεις που έχουν σχέση με την ε, κληρονομιά, διαδοχή κλπ. Ευχαριστώ. Και για την γλωσσική σας, το γλωσσικό σας κουράγιο. Προς το παρόν έχουμε ολοκληρώσει όλα τα σημεία της ε, ημέρησης διάταξης ε, που αφορούσαν τη δημόσια συζήτηση. Σε λίγο θα περάσουμε ε, σε εξέταση κάποιων σημείων και κλεισμένων των θυρών. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσουμε την συνάντησή μας αυτή μέχρι τις 5 η ώρα. Σας επιτρέπει να χαλαρώσετε λίγο.